επικυρώνεται η έγκριση. Από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, των Σοσιαλιστών, των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και την ΓΚΟΕ, έχω μια σειρά αιτούσεων για ορισμό μελών σε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και αντιπροσωπέ. Ο ελόγω κατάλογο θα ε, παρατηθεί στα πρακτικά τη τρέχουσα συνεδρίαση. Αν μέχρι την Έγκριση ε, στο πρακτικό δεν υπάρχει διαφωνία. Ισχύουν αυτοί οι ορισμοί. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων επίσης